Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, να επιστρέψουμε στις εργασίες μας. Φτάσαμε στο σημείο 11 που σημαίνει ότι θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μικ Βολέη που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, έχετε αναλάβει αυτή τη θέση από την αρχή της χρονιάς και σας καλούμε ε, στην Επιτροπή μας ε, για να, κάνουμε μια, να ξεκινήσουμε μια τακτική ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο της ΕΜΚΟ. Ο κάτοχός σας, ο Μπρούνο Κόκε, είχε έρθει, ο Μπρούνο Κόκε, είχε εδώ πέρσι και το περασμένο Μάρτιο είχαμε ανταλλάξει απόψεις με τον ε, εταίρο σας, θα τολμούσα να πω, της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας. Πριν σας δώσω το λόγο, θέλω να σας πω ότι επειδή έχουμε ξεκινήσει μια σχετικά νέα ε, πρακτική, τα μέλη δεν γνωρίζουν πολύ καλά το έργο και το ρόλο των επιτροπών αυτών που παρατάφτα γνωρίζουμε αποτελούν κάτι το πάρα πολύ χρήσιμο ε, από το, ένα χώρο από τον οποίο προέρχονται οι προτάσεις της Κομισιόν και που φτάνουν μέχρι το Συμβούλιο Υπουργών. Είναι ένα από τα όργανα του Συμβουλίου όπου τα κράτη-μέλη προετοιμάζουν τις ε, αποφάσεις με τη βοήθεια των εθνικών τους εμπειρογνωμόνων. Εν πάση περιπτώσει θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την δική σας πορεία και μετά να μας περιγράψετε ε, πώς έχουν τα πράγματα στην ΕΜΚΟ. Φυσικά γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο έχει κινητοποιηθεί λόγω της συζήτησης για το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης επί του οποίου έχουμε εκδώσει και γνωμοδότηση. Όμως είναι πολλά και τα υπόλοιπα θέματα επί των οποίων ε, έχουμε λόγο και βεβαίως μπορείτε και εσείς να συμμετάσχετε στη συζήτηση, να μας περιγράψετε πώς έχουν τα πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω ότι εδώ ξεκινά μια διαδικασία που θα συνεχιστεί. Η πρώτη συνεδρίασή μου ήταν ε, η την 1η Φεβρουαρίου, αλλά έκτοτε έχουν γίνει πολλά εντωμεταξύ. Μέχρι στιγμής παρακολουθούμε την ε, ετήσια έρευνα για την, ε, για την ανάπτυξη και επίσης συζητήσαμε την ε, έκθεση για την απασχόληση εν του Συμβουλίου ε, απασχόλησης είναι μία από τις δυνατότητες που έχουμε βάσει του άρθρου 148 της συνθήκης έχουμε την εξουσία αυτή. Επίσης παρακολουθήσαμε αυτή την πορεία αρκετά προσεκτικά εν του Συμβουλίου Απασχόλησης του Ιουνίου που επίκειται υπάρχουν διάφορα μέρη εδώ. Το ένα είναι πολύ καινούριο, είναι ένα παρατηρητήριο, μια παρακολούθηση των επιδόσεων που παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς ε, της επιδόσης των κρατών μελών λόγω του στόχου του 2020. Την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώσαμε την μελέτη των ε, NRPs, δηλαδή την, ε, ε, με, την έκθεση μεταξύ κρατών μελών του National Reform Program δηλαδή και βεβαίως θα συνεχίσουμε με τις ε, συστάσεις, με τις προτάσεις που φορούν κάθε κράτος μέλος και αυτή τη δυνατότητα την έχουμε νομοθετικά. Αναφερθήκατε στην Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά μαζί τους. Μιλάω με τον Λόρις ε, αρκετά συχνά και μου εξήγησε τα της επισκέψεώς του εδώ. Εκείνοι έκαναν ε, τη δική τους μελέτη των χωρών, των περιοχών του NRP, ε, που εμπίπτει στο δικό τους ε, χώρο. Μία Πέμπτη και Παρασκευή και Δευτέρα και Τρίτη συνεδριάσαμε και μαρθόμασταν δίπλα-δίπλα. Επίσης όλο και πιο συχνά συνεργαζόμαστε λόγω της φύσεως του 2020 με την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής η ΕΜΚΟ όμως με τα χαράς πρέπει να σας πω δεν ασχολείται με το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης. Είναι άλλοι που έχουν αυτή την ευθύνη. Χαίρομαι που εμείς δεν εμπλεκόμεθα. Χαιρόμαστε ε, με τη, για τη συνεργασία μας με τη, το EPC για τις διάφορες συστάσεις. Η Επιτροπή δηλαδή Οικονομικής, ε, την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής. μελετάμε τα θέματα τα πολιτικά και της πολιτικής. Επίσης, μόλις ολοκληρωθούν όλα αυτά και φτάσουμε επιτέλους καλοκαιρινές μας διακοπές, το φθινόπωρο θα δουλέψουμε για, σε κάτι νέο για μας. Είναι η θεματική παρακολούθηση όπου θα ασχοληθούμε πολύ λεπτομερέστερα σε, με κάποια βασικά θέματα μετά από τις ε, ε, μελέτες των NRPs που κάναμε, θέματα ας πούμε των ε, μεγαλύτερης ηλικία εργαζομένων, των ηλικιωμένων εργαζομένων ή τα θέματα των γυναικών κλπ. Τα κίτρινα και τα αντικίνητρα της αυξανόμενης συμμετοχής, όλα αυτά θα οδηγήσουν στη σύνταξη μιας έκθεσης για την ΕΠΣΚΟ του Δεκεμβρίου και μετά τα Χριστούγεννα θα ξαναρχίσει από την αρχή όλος αυτός ο κύκλος. Το... Τώρα, ποιο είναι το... Τι, καλύτερο... τι είναι το καλύτερο να κάνουμε, να περιμένω να μου κάνετε ερωτήσεις ή θέλετε κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσίαση. Α, α. Ε, θα αρχίσω πάλι να μιλάω γαλλικά, λέει η Πρόεδρος. Αντιλαμβάνομαι... Ε, ότι από τότε που αναλάβατε εσείς τα καθήκοντά σας το θέμα που κυριαρχεί είναι η παρακολούθηση αυτή του τρόπου με τρόπο που ακολουθεί το ευρωπαϊκό εξάμεινο και ουσιαστικά ε, το θέμα της απασχόλησης υπάρχει στο παράρτημα 3 της ετήσιας έρευνας για την ανάπτυξη. Είναι μια νέα εξέλιξη αυτή αν θέλετε και σημαντική μάλιστα. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι σε αυτή τη φάση στους διάφορους χώρους ευρωπαϊκής νομοθεσίας ε, υπάρχουν θέματα που, στα οποία πρέπει να μελετήσετε βαθύτερα. Θέλω να, να πω το εξής. Αυτά τα NRPs, τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης, σήμερα γίνεται μια πρώτη προσπάθεια. Είμαστε στην πρώτο έτος αυτού του κύκλου και θεωρώ ότι η Επιτροπή της οποίας προεδρεύεται έχει στη διάθεσή της όλα τα προγράμματα από όλα τα κράτη-μέλη. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να δουν τα μέλη τι πιστεύετε εσείς, ποια είναι η κρίση σας για την ποιότητα των ε, κειμένων που έστειλαν τα μέλη. Δεν ξέρω προηγουμένως με τι ασχολείστε ε, δηλαδή υπάρχει κάτι διαφορετικό τώρα, βλέπετε κάτι καινούριο σε αυτά τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης. Πώς λειτουργεί η Κομισιόν και κυρίως αυτή η μονάδα ε, παρά τη Γενική Γραμματεία της Κομισιόν με την ΕΚΦΗΝ και τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και πώς αξιολογείται και από απόψεως χρονοδιαγράμματος αλλά και από απόψεως περιεχομένου την όλη αυτή διαδικασία. Από άποψη χρονοδιαγράμματος εγώ από ό,τι κατάλαβα υπάρχουν κάποια σημαντικά βήματα. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις ε, έχουν πάρα πολύ πιεστικές προθεσμίες. Πώς έχει ξεκινήσει όλο αυτό, είναι κάτι το καθαρά τυπικό ή υπάρχει δυνατότητα επηρεασμού ε, της κατάστασης και επί της ουσίας ε, ποια είναι η συζήτηση, ποια είναι η φύση της συζήτησης γιατί πολλά είναι τα στοιχεία της έκθεσης για την ετήσια ανάπτυξη που μπορούν να ε, επισύρουν κριτική όπως το θέμα της ε, ηλικίας συνταξιοδότησης, ε, το θέμα της μεταρρύθμισης των μισθών κλπ. κλπ. Αυτό συζητείτε στην Επιτροπή σας, στην ΕΜΚΟ. Και με ποιο τρόπο, πώς. Θα σας αφήσω να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα τώρα και μετά ίσως να, αφήσουμε, να δώσουμε το λόγο και στους άλλους συναδέλφους. Uh, Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι συνεκτικός και να μην μακρηγορήσω για να έχουν χρόνο και συνάδελφοι να θέσουν ερωτήσεις. Καταρχήν, στην εξέταση ε, των διαφόρων χωρών, στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, ε, η δουλειά οργανώνεται σε workshops. Γίνονται συναντήσεις ομάδων κρατών μελών και στη συνέχεια συνεδριάζουμε ξανά σε Ολομέλεια για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα. Σε αυτές τις ομάδες κρατών μελών μία χώρα αρχίζει να συζητάει θέματα με άλλες χώρες, ε, υποβάλλουν κάποια ζητήματα προς αξιολόγηση, πράγμα το οποίο κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορούμε να δούμε και τις δύο πλευρές και τις δύο απόψεις των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή. Αυτή τη φορά είδαμε ότι ε, υπήρχαν κοινά σημεία σε αυτά τα οποία συζητούσε η Επιτροπή και αυτά που συζητούσαν τα κράτη-μέλη, αν και υπήρχαν και κάποιες διαφορές. Προσπαθούμε να έχουμε χρόνο για συζήτηση και όπως είπατε και εσείς είναι ο πρώτος χρόνος των νέων εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης σύμφωνα με τη νέα στρατηγική για το 2020 άρα η αξιολόγηση δεν αναμένεται να είναι τόσο πλήρης και λεπτομερής ε, όσο θα περίμενε κανείς. Γιατί πολλά κράτη-μέλη προσπαθούν να δουν ε, τον ορίζοντα των 10 ετών, άλλα κράτη-μέλη προσπαθούν να τα κάνουν όλα στην αρχή, ενώ άλλα τα αφήνουν περισσότερο για το βάθος ε, των 10 χρόνων. Συζητάμε λοιπόν τις πιθανές αξιολογήσεις χωρίς να έχουμε ακόμη συμπεράσματα και πρόκειται να πούμε στους υπουργούς ποιες είναι οι προκλήσεις και τι χρειάζεται να γίνει γιατί προς το παρόν δεν μπορούμε να έχουμε τελικά συμπεράσματα. αυτό είναι ένας από τους λόγους ε, για τη νέα αυτή επιτήρηση, τον, νέα αυτή εποπτεία των διαφόρων θεμάτων για να μπορέσουμε να έχουμε μια γενικότερη εικόνα αναθέμα και αναχώρα. Ε, και το θέμα της ενεργού ε, ζωής και τη επέκταση του χρόνου εργασία για του ηλικιωμένου εργαζομένου, είναι ένα από τα θέματα που συζητάμε, όπω και άλλα θέματα, όπω φορολογικά κίνητρα, το ευρύτερο θέμα των συνθήκων εργασία, υποστήριξη ε, από τον εργοδότη κλπ. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, η πίεση που υπάρχει αφορά τις συστάσεις, γιατί στις 7 Ιουνίου θα δημοσιεύσει μια δέσμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα θέματα που αφορούν την απασχόληση έχουμε στις 17 Ιουνίου το Συμβούλιο των Υπουργών Απασχόλησης. Αν βγάλετε λοιπόν και τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες βλέπετε ότι μας μένει πολύ λίγος χρόνος. Γι' αυτό υπάρχει πίεση. Πίεση προς όλους και στα κράτη-μέλη και στην Επιτροπή και ε, στις ομάδες του Συμβουλίου και της Προεδρίας. Ελπίζω ότι θα έχουμε το χρόνο να το σκεφτούμε για να δούμε πώς τις επόμενες χρονιές μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή τη διαδικασία που τώρα εφαρμόζουμε για πρώτη φορά. Και θα προσπαθήσουμε και κατά τα επόμενα έτη να κάνουμε μια εις βάθος εξέταση και μια συζήτηση που θα ασκεί σε βάθος κριτική στα διάφορα θέματα. Τώρα είναι ακόμη πρώτος χρόνος και πολύ νωρίς για να δούμε κάποια από τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γούλη για την, ε, για την ενημέρωση που μας κάνατε και για όλα όσα μας είπατε, τα οποία τροφοδοτούν, αν θέλετε, τη γενικότερη συζήτηση. Για να σας ξεκαθαρίσω τα πράγματα, να σας πω ότι είμαι και λίγο σκεπτικιστής σε σχέση με αυτά που μας είπατε. Είμαι Ισπανός. Στην Ισπανία το 50% των νέων είναι άνεργοι. Ε, χιλιάδες άτομα έχουν καταλάβει τις πλατείες ε, ε, της χώρας μας. μας. Και οι τις οποίες δίνει η Ευρώπη, είτε είναι από την Κομισιό, είτε είναι από το Κοινοβούλιο, πόρο απέχουν ε, από το να δείξουν μια ευαισθητοποίηση για, τα, για την κατάσταση που βρίσκονται τα άτομα αυτά. Του ζητάμε να προσαρμοστούν εκείνοι σε ένα τρελό οικονομικό σύστημα το οποίο δεν προσφέρει καμία απάντηση στις ανάγκες τους. Κύριε Γούλε, η Επιτροπή σας αποτελείται από έντιμους ε, ε, ειδικού. Αλλά να ρωτήσω, μήπως η όλη διαδικασία είναι πολύ γραφειοκρατική, λαμβάνοντας υπόψη ε, την, τον επίγοντα χαρακτήρα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι, οι πολίτες της, της Ένωσης. Ένα αυτό. Δεύτερον, βλέποντας τι γίνεται στα διάφορα συμβούλια Υπουργών Οικονομικών κτλ, βλέπουμε ότι η Ευρώπη ε, αναλαμβάνει δράση ε, εναντίον αυτών που δεν σέβονται κάποιες ε, παραμέτρους, ε, κάποιες ε, υποχρεώσεις κτλ. Και όντως όλοι κάνουν κάποιες προσπάθειες, είτε είναι το Συμβούλιο είτε είναι οι Υπουργοί. Αλλά διερωτώ με μήπως θα έπρεπε το Συμβούλιο να παρουσιάσει, να, να, να εξετάσει λίγο παραπάνω τα όσα γίνονται στον τομέα της απασχόλησης, να δούμε από κοντά ποια είναι η κατάσταση, ποιο είναι το δικαίωμα εγκατάστασης κτλ. Επίσης αναφερθήκατε στις συνέπειες των προγραμμάτων προσαρμογής, ε, δημοσιονομικής προσαρμογής στο, στην απασχόληση. Υπάρχουν τα, υπάρχει το χρέος, το, το δημόσιο χρέος κάποιων κρατών. Ε, δεν υπάρχουν ε, δυνατότητες ε, το κράτος να καλύψει την έλλειψη ιδιωτικών πρωτοβουλειών. Οπότε ρωτώ, έχετε εσείς κανένα, κάποια πληροφορία για τον αντίκτυπο που έχουν τα προγράμματα προσαρμογής του Συμβουλίου. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Μία γενική απάντηση στο γενικότερό σας ε, ερώτημα είναι για το κατά πόσο η Επιτροπή Απασχόλησης θα εξετάσει ε, πακέτα προσαρμογής, ε, πακέτα δημοσ... ολοκλήρωσης της δημοσιονομικής πολιτικής κτλ. Η απάντηση σφαιρικά είναι όχι, διότι όλα αυτά τα πακέτα ανήκουν στην αρμοδιότητα των Υπουργών Οικονομικών. Όμως, όπως σας είπα, θέλουμε να συνεργαστούμε κοντά με την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής και συνομιλώ με τον πρόεδρό τους αυτή τη στιγμή για να δούμε τι κοινή δουλειά μπορούμε να κάνουμε. Επίσης, δεν επικράτησε σιωπή, αν θέλετε, για τα θέματα αυτά. Συζητήθηκαν αλλά δεν κρίνουμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων πακέτων. Θα το συζητήσουμε, ε, εξετάζουμε τα, τις συνέπειες στην απασχόληση στην, τις συνέπειες στην απασχόληση, γιατί θα το συζητήσουμε και με τους υπουργούς ε, τι πολιτικές πρέπει να εφαρμόσουμε ε, για να παρουσιαστεί μια κάποια, προκαλέσουμε κάποια ανάκαμψη στον τομέα της απασχόλησης. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσουμε ε, λαμβάνοντας υπόψη ε, και τα, τις κοινωνικές πτυχές ε, ότι οι άνθρωποι που αξίζουν δεν θα μείνουν απ' έξω είναι σίγουρο ότι η κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί πριν από την, από την κρίση δεν είχε βοηθήσει και όλους στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτή η γενικότερη κρίση, η γενικότερη αξιολόγηση την οποία ε, εσείς θα θέλατε. Ε, αλλού θα πρέπει να γίνει αυτό. Ένα άλλο θέμα χωρίς να διαφωνώ με τίποτα από αυτά που είπατε. Ε, δεν νομίζω ότι ούτε η Ισπανική κυβέρνηση, ούτε ο, Ισπανός, ε, ο Ισπανικός λαός περιμένει την Επιτροπή Απασχόλησης ε, για να τους, για να τους δώσει μια λύση. Η κυβέρνηση της Ισπανίας προσπαθεί, οι πολίτες της Ισπανίας με την ψήφο τους δίνουν την απάντησή τους ε, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη δουλειά. Εμείς σαν Επιτροπή Απασχόλησης ε, ε, δεν μπορούμε να αναδιαρθρώσουμε πλήρως και εκ βάθρων μια πολιτική, την πολιτική απασχόληση μιας χώρας. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω, από το 1997 πολλά πράγματα έχουν ε, αλλάξει, έχουν βελτιωθεί, υπάρχει διαδικασία του Λουξεμβούργου, ε, υπάρχουν αυξημένα επίπεδα συμμετοχής, βέβαια τα αποτελέσματα, όπως είπατε και εσείς, τα αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 2010 δεν ήταν ε, τα αναμενόμενα, ήταν τα επιθυμητά. Ο συντονισμός και η συνεργασία παρουσιάζει κάποια αποτελέσματα, όμως δεν είναι αυτό που θα μας λύσει όλα τα προβλήματα. Δεν ξέρω αν ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε αυτή η ευκαιρία να συζητήσουμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση ε, στην οποία ε, έχουμε ανάπτυξη χωρίς να έχουμε αύξηση της απασχόλησης. Η ομάδα εργασίας σας ε, ασχολείται με τις διάφορες τάσεις της απασχόλησης με το τι συμβαίνει δηλαδή μέσα στην απασχόληση, αν υπάρχουν κάποιες νέες τάσεις, κάποιες ορατές τάσεις στη δομή της απασχόλησης. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να βελτιωθεί ώστε να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό στον τομέα της απασχόλησης. Ο κύριος Γουλή. Ευχαριστώ. Αλλά ε, ήθελα να υπενθυμίσω και ε, όσον αφορά την ερώτηση προηγουμένως για το τι μέτρα παίρνει αυτή η Επιτροπή υπάρχουν ε, οι συστάσεις τις οποίες κάνουμε απευθείας προς τα κράτη-μέλη αυτό ξέχασα να το αναφέρω τώρα για την ερώτηση της ε, κυρίας Μπάουερ Υπάρχει και άλλη μια επιτροπή με τους εμπειρογνώμονες που ασχολούνται ακριβώς με τα θέματα αυτά. Εμείς βεβαίως ανταλλάσσουμε απόψεις με την Επιτροπή εκείνη και έχουμε άποψη για το πώς θα μπορούσε μακροπρόθεσμα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να είναι αποτελεσματικότερο. Δεν θα ήθελα να μιλήσω εγώ καθαρά για το κοινωνικό ταμείο, αν και συνεργαζόμαστε με αυτό το θέμα. Για την πρώτη σας ερώτηση τώρα για την ανάπτυξη χωρίς απασχόληση, αυτό είναι ένα από τα βασικά μελήματα της Επιτροπής Απασχόλησης και του Συμβουλίου και το έχουμε επισημάνει και στα συμπεράσματα. Την Πέμπτη και την Παρασκευή κατά την τρέχουσα εβδομάδα έχουμε δύο συνεδριάσεις και στη μία από τις δύο οπωσδήποτε θα συζητήσουμε το τι μπορεί να κάνει η απασχόληση, ε, τι μπορούν να κάνουν οι Υπουργοί Εργασίας και Απασχόλησης για να βελτιώσουν και την ε, πλευρά ε, της ε, προσφοράς και την μακροπρόθεσμη κατάσταση των, ε, των εργαζομένων και των μακροπρόθεσμα ανέργων. Είναι προκλήσεις πολύ πιεστικέ, τις οποίες θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και εκτός από την πλευρά της προσφοράς θέλουμε να δούμε και την, την πλευρά της ζήτησης, πώς μπορούμε δηλαδή ε, να δώσουμε κίνητρα στους εργοδότες, πώς μπορούμε ε, να ε, κάνουμε τους εργοδότες να απασχολήσουν περισσότερους ε, ανέργους. Είναι θέματα τα οποία ε, ετοιμάζουμε και στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης που ανέφερα προηγουμένως και τα θέματα που γενικότερα μας απασχολούν. Και για το θέμα των ορών εργασίας, ε, θέλω να σας πω ότι είναι ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούν. Οι εταιρείες συνεχίζουν να μετατρέπουν ε, τις ε, ε, σχέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης σε σχέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, κάτι το οποίο υπήρχε στο παρελθόν και είναι και αυτό ένα από τα θέματα που απασχολούν την Επιτροπή μας. Ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Θα ήθελα να επανέλθω de votre intervention dans l'ensemble Λοιπόν, μα έκανε ιδιαίτερη εντύπωση κατά τη διάρκεια της Βελγική προεδρία η κινητοποίηση που είχε οργανώσει η Βελγική Προεδρία για να έχει στη διάθεση της η ΕΠΣΚΟ, η Επιτροπή δηλαδή, η, ε, Επιτροπή, ε, κάποιες ε, ε, κάποιους δείκτες, ε, κάποιες πληροφορίες ε, για να μπορεί να συνομιλήσει με το ΕΚΟΦΗΝ. Και ο προκάτοχός σας, από ό,τι θυμάμαι, έλεγε ότι το να έχει η Επιτροπή στη διάθεσή της ένα ολόκληρο οπλοστάσιο δικτών και συντελεστών κτλ. ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, εσείς τι έχετε κάνει για το θέμα αυτό, έχετε προχωρήσει και ξέρω ότι είσαστε και μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων της ΕΠΣΚΟ. Αλλά όταν ε, το εγχειρίδιο δημοσιεύθηκε, ε, προκάλεσε κριτική, κυρίως όσον αφορά το περιεχόμενό του στο κοινωνικό τομέα. Και για τον τρόπο με τον οποίο φαινόταν να παρακάμπτει τις πρακτικές και τις ανάγκες κοινωνικού διαλόγου. Λοιπόν, να συζητήσεις για να προετοιμάσει, προετοιμαστεί η ΕΠΚΟ στο σημείο αυτό. Κοιτάξτε. Το θέμα των δικτών συμφωνώ με αυτό που σας είπε ο Μπρούνο και ανέφερα εν συντομία ε, αυτό το θέμα της, ε, των ε, δικτών επίδοσης ή απόδοσης. Θα στηρίζεται σε μία σειρά δικτών που θα προέρχονται, που θα συλλέγονται μακροπρόθεσμα. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή και η προσπάθεια αυτή θα γίνει ε, μέσα στα πλαίσια ενός προγράμματος ε, στο οποίο συμμετέχει και η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Βέβαια, μέσα στα πλαίσια της ύφεσης, όταν παρουσίασε η ύφεση, όντως αντιδράσαμε εκ των υστέρων αλλά το φθινόπωρο θα έχουμε μία έκθεση η οποία θα υποβληθεί ε, το Δεκέμβριο στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και θα δημοσιευθεί πριν από την ετήσια ε, ε, τον τίσιο την τήσια μελέτη ε, για την ανάπτυξη. Αυτή είναι η συνεισφορά, η μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς στον τομέα της ανεργίας και της κοινωνικής πολιτικής πριν να βοηθήσουμε την Κομισιόν δηλαδή, πριν την δημοσίευση του πακέτου της στην Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας θα υπάρξει και μια έκθεση που θα αφορά την δική τους διάσταση, την κοινωνική διάσταση στα θέματα φτώχειας και αποκλεισμού. Επομένως, αν όλα πάνε καλά, το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης θα είναι το πρώτο το οποίο θα έχει στη διάθεσή του όλα αυτά τα θέματα και θα μπορέσει να, να μιλήσει για τα θέματα απασχόλησης. Μια συμπληρωματική ερώτηση, μια και έχουμε χρόνο. Στα κείμενα, τα νομοθετικά κείμενα, τα οποία συζητάμε εδώ, στην Επιτροπή Απασχόλησης, υπάρχει η οδηγία για τον χρόνο απασχόλησης, οδηγία για την οποία, την οποία ε, συζητήσαμε και ψηφίσαμε στην προηγούμενη θητεία κλήθηκαν αρκετές συζητήσεις ε, λόγω της συμμετοχής και των κοινωνικών εταίρων προσπαθήσαμε να βρούμε μια συμφωνία πάνω σε αυτή την οδηγία. Επομένως εσείς ε, στην ΕΜΚΟ το θίξατε το θέμα ή είναι νωρίς ακόμα στα πλαίσια της διαδικασίας σας και περιμένετε μια πρόταση της Κομισιόν για να το συζητήσετε. Μια ερώτηση αυτή και δεύτερη. Στο πακέτο οικονομική διακυβέρνηση υπάρχει μια πρόταση που αυτή τη στιγμή δεν είναι επιτάπητος μένα, αλλά που συζητάτε συχνά στους διαδρόμους, είναι ο μηχανισμός κυρώσεων που θα ε, δημιουργηθεί, που θα πρέπει να ερμηνευθεί σαν μία μείωση των χρημάτων, των ποσών που χορηγούνται στα κράτη-μέλη μέσα στα πλαίσια και ενδυνάμει μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είχατε τη δυνατότητα να το συζητήσετε αυτό το θέμα και αν ναι, πώς μπορείτε να επηρεάσετε την κατάσταση. Yes, And I should apologize you. Ναι, θίξατε το θέμα αυτό και την προηγούμενη φορά ε, δεν το δεν απήντησα. Επανήλθα, λέει η κυρία Περές. Ναι, ζητώ συγγνώμη, λέει ο κύριος Γούλη. Θα απαντήσω τώρα. Δεν θα συζητήσουμε όμως, δεν συζητάμε την νομοθεσία εμείς. Εμείς σαν Επιτροπή Απασχόλησης δεν έχουμε τέτοιου είδου αρμοδιότητα. Οι ομάδε εργασία και η Επιτροπή και διάφορες επιτροπές άλλες ε, ασχολούνται με το θέμα αυτό. Ο ρόλος της Επιτροπής Απασχόλησης αναφέρεται στο άρθρο 148 και αφορά τη διαδικασία Λουξεμβούργου. Είναι η στρατηγική, η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, αν το θυμόσαστε. Και δεν, είναι, δεν έχει νομοθετικό περιεχόμενο. Όμως θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχει και ένας διάλογος ο οποίος εντείνεται με την ε, Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής, με την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και αυτό μας έχει προσεγγίσει περισσότερο με τους κοινωνικούς εταίρους. Τους ε, ε, συναντήσαμε επίσημα τρεις φορές φέτος και συζητήσαμε ε, την ε, κοινή έκθεση για την απασχόληση, συζητήσαμε κάπως, είδαμε τα εθνικά προγράμματα και ελπίζουμε ότι θα συναντηθούμε εκ νέου και θα συζητήσουμε όλα τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν και το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης το Δεκέμβριο. Επομένως, όπως σας είπα θα κάνουμε εμείς και τις δικές μας δηλώσεις πριν από την ε, ε, ε, επόμενη ετήσια έκθεση για την απασχόληση. Για την ανάπτυξη, συγγνώμη. Πάντως, ουσιαστικά, εμείς δεν παίζουμε κανένα ρόλο σε, σε καμία πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Δεν έχουμε να κάνουμε με την, με την νομοθεσία. Τώρα, ε, για το, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει μια τεχνική επιτροπή. Θίξατε όμως ένα θέμα που μου έφερε μια ιδέα. Θα πρέπει να δούμε πώς η Επιτροπή Απασχόλησης μπορεί να γνωμοδοτεί ή να δώσει κάποια άποψη, κάποια συμβουλή για, τον, για την λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ούτω ή άλλω την επόμενη περίοδο θα αναδιαρθρωθεί η λειτουργία του. Ε, εξού και θα το σημειώσω και θα το συζητήσω με την Επιτροπή πολύ καλά. Λοιπόν, συγχαρητήρια ε, γιατί το πέρασμά σας από εδώ τροφοδότησε το πρόγραμμα εργασίας μας ως Επιτροπή Απασχόλησης. Από ό,τι βλέπω δεν θέλει κάποιος να πάρει το λόγο, οπότε μπορούμε να σας ευχαριστήσουμε και να κλείσουμε ραντεβού μαζί σας ε, για μια άλλη ε, συζήτηση που θα επαναλαμβάνετε τακτικά. Και μην διστάσετε αν την οποιαδήποτε στιγμή ε, θέλετε κάποια να πάρετε τον λόγο, να παρέμβετε, να έρθετε σε επαφή με τα μέλη της Επιτροπής. Μην διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθειά μας. Πάντα έχουμε χρόνο για τέτοιου είδους ε, επαφές. Ευχαριστώ. Très bien. Πάρα πολύ ωραία. Η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε προγραμματίσει ολοκληρώθηκε ταχύτερα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια του σημείου 12, τη Ρεγκίνα Πάστος, που μπόρεσε ήδη να βρίσκεται εδώ. Θα της δώσω το λόγο για να συζητήσουμε το σχέδιο εκθέσης της που ε, αφορά μία από τις σοβαρές πρωτοβουλίες της ε, Επιτροπής και τα θέματα που την απασχολούν την ατζέντα για τις νέες δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας. Agenda for New Skills and Jobs. Κυρία εισηγήτρια, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Φυσικά θα είστε η εισηγήτρια επί της ουσίας και εμείς θα έχουμε γνωμοδοτήσεις από τις Επιτροπές Ήτρε, Ρεζή, ε, Πολιτισμού και Γυναικών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, είναι προνόμιο για μένα που μου δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσω την έκθεση για το εξαιρετικά σημαντικό αυτό θέμα που αφορά τις νέες δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας στα πλαίσια μιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που επηρεάζει και πλήττει την Ήπειρό μας. Βρισκόμαστε σε, μια περίοδο ε, αυξημένης ανεργίας 23% ε, οι νέοι ε, έχουν ανεργία σε επίπεδο 21% και έχει συνεχή αύξηση η μακροχρόνια ανεργία. Αυτό βεβαίως έχει σοβαρές συνέπειες για τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και δημιουργεί θεμελιώδη προβλήματα. Η δημιουργία θέσεων εργασίας και η δυσκολία εξέβρεσης ατόμων που έχουν ε, τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις ε, προσφορά εργασίας είναι η κατάσταση. Οπότε μας παρουσίασε η Κομισιόν την ανακοίνωση για την ατζέντα για τις νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας ε, ε, που παρουσιάστηκε σε εμά τον περασμένο Νοέμβριο στο Στρασβούργο, σχετικά πρόσφατα δηλαδή. Η ατζέντα είναι με δύο λόγια η στρατηγική του 2020 υπέρ μιας έξυπνης βιώσιμης ε, ανάπτυξης, ε, δηλαδή μια σειρά από εφημισμούς που ακούγαμε μέχρι τώρα διαρκώς. Η Κομισιόν προσπαθεί να συνεισφέρει στην αύξηση ε, της απασχόλησης των Ευρωπαίων πολιτών θέλουμε 75% των ανθρώπων πάνω από το 64% που θα θέλουμε να δουλεύουν μέχρι το 2020. Υπάρχει δυνατότητα, σημαντική δυνατότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, είτε νέων είτε άλλων ε, συμπληρωματικών σε πολλούς χώρους, στην ε, τεχνολογία αλλά και στον χώρο παροχής υπηρεσιών. Το δεύτερο συμπέρασμα της Κομισιόν είναι ότι οι ανάγκες όσον αφορά τα προσόντα αυξάνονται σημαντικά. Για πάσης, για κάθε είδους ε, ε, επάγγελμα σε κάθε επίπεδο. Πρέπει οι υποψήφοι να είναι πιο μορφωμένοι πολύ σύντομα και θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αντιστοιχία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Θεωρούμε ότι είναι σωστή η προσέγγιση αυτή της Κομισιόν. Μας ε, Βρίσκουμε πολύ ενδιαφέρουσα την ανάλυση της ΣΕΦΕΤΟΚ. Γίνεται μια ανάλυση των αναγκών και αναφέρονται τέσσερις βασικοί τομείς προτεραιότητες. Η αγορά, η αγορά εργασίας, οι δεξιότητες και οι πολιτικές θα στοχεύουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ε, τι στοχεύουμε στο σχέδιο έκθεσης αυτό. Να είμαστε πιο συνοπτικοί Ξέρουμε ότι υπάρχουν όρια Α. Ε, λοιπόν, λαμβάνω, ε, λαμβα, αν λάβουμε όλα αυτά υπόψη, θεωρώ ότι έχουμε συμπεριλάβει τα πιο σημαντικά όσον αφορά το μέλλον, δηλαδή ότι καταρχάς θα χρειαστούμε ε, περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό στο μέλλον. Μέχρι το 2020 οι θέσεις ε, απασχόλησης ε, θα που χρειάζονται υψηλά προσόντα θα είναι από 25% σε 31%. Για τα μεσαία προσόντα θα υπάρχει μία μικρή αύξηση και θα υπάρχει επίσης και ένα ποσοστό θέσεων απασχόλησης που δεν χρειάζονται ιδιαίτερα προσόντα και το ποσοστό αυτό από 26% που είναι τώρα θα φτάσει στο 18%. Θα, στην, Ευρώπη των 25 έχουμε 6 Έχουμε 6 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης 6 ε, εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια ε, νέες θέσεις απασχόλησης και ένα μεγάλο μέρος, ένα μεγάλο ποσοστό των θέσεων αυτό είναι ε, εξειδικευμένοι εργαζόμενοι. Άρα υπάρχει μια πρόκληση την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τώρα όσον αφορά την μετανάστευση, ε, όλες αυτές οι, όλα αυτά τα μεταναστευτικά ρεύματα, οι μεταναστευτικές ροές θα επηρεάσουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη μας ε, και την πράσινη οικονομία η οποία θα επηρεάσει πάρα πολύ τον τομέα της απασχόλησης στην, ε, στην ανακύκλωση, στην, στις μεταφορές, στην ενέργεια. Υπάρχουν, υπάρχουν όλες αυτές οι προκλήσεις που θέλουμε να έχουμε μια βιώσιμη, μια οικολογική οικονομία. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε τους ανθρώπινους πόρους μας να αποκτήσουν νέες ικανότητες, νέα προϊόντα, νέα προσόντα η Ευρώπη θα ε, παράγει νέα προϊόντα, ε, καινοτόμα προϊόντα και θα πρέπει να βοηθήσει τους εργαζόμενους να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα. Ένα άλλο, μια άλλη πρόκληση αν θέλετε αφορά τους νέους. Χρειάζονται ε, μέτρα έτσι ώστε να περιοριστεί η η φυγή από το σχολείο ε, είναι και, αυτή, και αυτός ένας από τους στόχους ε, της πολιτικής της στρατηγικής μας για το 2020. Επίσης θα πρέπει να εναρμονίσουμε κατά τον τρόπο αναγνώρισης ε, των προσόντων έτσι ώστε να διευκολύνουμε την μετακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διότι εκεί είναι ο μεγάλος όγκος και των θέσεων απασχόλησης αλλά και της ανεργίας. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις ε, επενδύσεις που θα χρειαστούν ε, στο μέλλον για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια συνεργασία με τα κέντρα εκπαίδευσης και για την ε, επιμόρφωση, των, κατάρτιση των ε, εργαζομένων, αλλά και για την διαβίου μάθηση. Ελπίζω ότι ανέφερα τα πιο βασικά στοιχεία αυτής της ε, έκθεσης. Στηρίζομαι στη συνεργασία όλων και τις 15 Ιουνίου θα υπάρχει μία ακρόαση, δημόσια ακρόαση για τους και με τους εμπειρογνώμονες. Πιστεύω ότι αυτό θα ε, βοηθήσει γιατί θα δούμε ποιες είναι οι προοπτικές στον τομέα αυτό και περιμένω και την, ε, τις νομοδοτήσεις των άλλων δύο επιτροπών που ε, θα βοηθήσουν στην ολοκλήρωση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Monsieur Puis... Ο Σερκάς, και η κυρία Σούτερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η σκιώδης εισηγήτρια, η κυρία Ρεσβάνα Πλάν, θα έρθει από στιγμή σε στιγμή. Έπρεπε να, βρίσκεται, να βρίσκεται σε άλλη συνεδρίαση. Θα ήθελα όμως να πω δύο λόγια εκ μέρους της πριν έρθει εδώ. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Ρεγκίνα Πάστος για το σχέδιο έκθεσης που συνέταξε. Σε γενικές γραμμές το θεωρούμε σημαντικό ένα έγγραφο, ένα κείμενο που λαμβάνει υπόψη του τις νέες ευκαιρίες που μπορούμε να ε, εντοπίσουμε και εμείς τη νέα αυτή εμβληματική πρωτοβουλία. Όπως σας είπα το έγγραφο για μας, το κείμενο αυτό είναι σημαντικό, είναι απαραίτητο ε, καθώς προχωρούμε στο μέλλον, όπου πρέπει να ανοίξουμε σε νέες θέσεις εργασίας και σε νέες δεξιότητες. Αυτό είναι απαραίτητο. Αν δείτε τις χώρες μας υπάρχουν θέσεις εργασίας ξεπερασμένες που πρέπει να αλλάξουν και να μεταρρυθμιστούν. Το θέμα είναι πολύ σύνθετο. Θέλω όμως να επισημάνω τρία ε, ε, θέματα που θα θέλαμε να, να τύχουν περαιτέρω επεξεργασία στο σχέδιο αυτό έκθεσης. Καταρχήν το θέμα αυτό της flexicurity. Αν ε, μελετήσετε την παράγραφο 6 ε, για να ε, απλουστεύσουμε τα πράγματα, η πολιτική μας ομάδα είναι διατεθειμένη να συζητήσει για το flexicurity. Μην ξεχνάμε όμως ότι αυτό το μοντέλο προέρχεται από εξαιρετικά ανεπτυγμένες χώρες με τεράστια δυνατότητα για επενδύσεις και πρόκειται για μια και που έχουν μια δομή που δεν αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα όπως ε, αντιμετωπίζουν κάποιες άλλες χώρες. Αν λοιπόν πάρουμε το μοντέλο flexicurity και ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών διαφόρων χωρών, την, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που υπάρχουν εκεί. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να ε, εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο flexicurity σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν χώρες που δεν θα μπορέσουν να εξισορροπήσουν τη flexicurity την, ευελιξία και την ασφάλεια της θέσης εργασίας. Ε, εδώ πρέπει δηλαδή να αναφερθεί και μια διάγνωση στο κείμενο. Δεν θα πρέπει δηλαδή αυτή η flexicurity να αναφέρεται με τόσο απόλυτο τρόπο. Δηλαδή δεν πρόκειται για μια πανάκια που θα λύσει παν πρόβλημα. Ε, ε, είναι ένα θέμα που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Πρέπει επίσης να μπορέσουμε να σεβαστούμε την απαραίτητη δημοσιονομική πειθαρχία. Αλλά δεν είναι το ίδιο να το εφαρμόζει αυτό, αυτό κανείς τα τρέχοντα έξοδα του δημοσίου τομέα σε πάρα πολλές χώρες πρέπει να αυξηθεί η απασχόληση, να αυξηθεί η δραστηριότητα της οικονομίας. Η Ρεγκίνα Μπάστος αντιμετωπίζει κάπως μονόπλευρα το θέμα γιατί επικεντρώνεται στη δημοσιονομική πειραθία που επαναλαμβάνω είναι σημαντική αλλά τι θα γίνει με τα επενδυτικά προγράμματα, τα προγράμματα που θα δώσουν μια ε, ε, ε, νέα όθηση στην οικονομία. Και τέλος κυρία Πρόεδρε, το ανέφερε και η Ρεγκίνα, αλλά όσον αφορά την ομάδα μας, η εκπαίδευση και οι ίσες ευκαιρίες είναι σημαντικές. Αν θέλουμε όμως την εκπαίδευση και τις ίσες ευκαιρίες για όλους, δεν θα πρέπει να αφήσουμε το θέμα ε, στην αγορά υπάρχουν κάποιοι που δυσκολεύονται περισσότερο να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε δημόσια παιδεία, παιδεία που να επικεντρώνεται στα λιγότερα ευνοημένα μέλη της κοινωνίας και προσφέρει ίσε ευκαιρίες για να είναι πραγματικές ίσες ευκαιρίες, να μην μένουν μόνο στα λόγια ε, ε, θα πρέπει να μην περιοριστόμαστε μόνο ε, στις πρωτοβουλίες της αγοράς. Δεν θα τις δημιουργήσει η αγορά. Χρειάζονται χρήματα. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα χρήματα δεν θα μπορέσουν να αγοράσουν αυτού του είδους την παιδεία. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρουμε μερικές ιδέες που είναι συμπληρωματικές σε αυτές που έχουν ήδη διατυπωθεί. Κύριε Σουέτερ. θα πρέπει να δώσω δίκαιο στην άλφα Σέρκα σε πολλά θέματα. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαμε πολλές ελπίδες ότι αυτή η ανακοίνωση ε, θα κάλυπτε σε μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις δυνατότητες για απασχόληση, για τις δυνατότητες σε μια ε, νέα ε, κοινωνία με ανάπτυξη της απασχόλησης. Αυτά περιμέναμε από την Επιτροπή. Όταν δούμε όμως αυτή την ανακοίνωση της Επιτροπής, ε, θέτει αλλού τη βαρύτητα η Επιτροπή. Θέτει τη βαρύτητα στις ευέλικτες αγορές εργασίας και δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ε, αν θέτει μάλιστα τη βαρύτητα στο ε, να εκλείψουν κάποια από τα βασικά ε, θέματα της προστασίας της αγοράς εργασίας. Δεν ανταποκρίνεται λοιπόν στις προσδοκίες μας αυτή η ανακοίνωση και δεν ανταποκρίνεται και στις προσδοκίες των πολιτών, στην Ισπανία ιδίως και βλέπουμε τώρα πώς ξεσηκώνονται οι νέοι στην Ισπανία και λένε ότι θέλουν μια νέα πολιτική απασχόλησης. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με αυτό το οποίο παρουσιάζει η Επιτροπή, τουλάχιστον με το πρώτο τμήμα. Και εδώ η συγγήτρια καλύπτει σωστά αυτό τον τομέα, γιατί θέλουμε νέες δεξιότητες για νέε θέσεις απασχόλησης και έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει να δούμε πού υπάρχουν ανάγκες κατάρτισης, τι πρέπει να κάνουμε για να ανταποκριθούμε στην πρόκληση ε, της νέας οικονομίας ε, και των νέων δεξιοτήτων και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό. Και ε, αυτή την έκθεση θα ήθελα σε αυτά τα βασικά σημεία να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Το θέμα του τι σημαίνει η εκπαίδευση και ευελιξία σε σχέση με τις θέσεις απασχόλησης δεν νομίζω ότι το χρειαζόμαστε σε μια τέτοια γνωμοδότηση. Έχουμε συζητήσει τα θέματα της ευελιξίας, έχουμε συζητήσει τα θέματα κατάρτισης μέσα την ε, ε, απασχόληση και ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, αλλά εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται προς άλλη κατεύθυνση σε διαφορετικούς τομείς από ό,τι εμείς είχαμε ελπίσει ότι θα έχουμε σε μια τέτοια γνωμοδότηση, σε μια τέτοια ανακοίνωση, ούτε ώστε και η δική μας γνωμοδότηση να καλύπτει θέματα ε, του εργατικού δικαίου κλπ. Τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά και πιστεύω ότι η βαρύτητα πρέπει να τεθεί σε άλλα σημεία. Ήδη στο Κοινοβούλιο έχουμε ε, εκφράσει τις απόψεις μας για το θέμα αυτό σε προηγούμενε γνωμοδοτήσει και σε κάτι τέτοιο θα έπρεπε να ανταποκρίνεται η ανακοίνωση της Επιτροπής. Θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις στους νέους, στους νέους που βρίσκονται στους δρόμους της Μαδρίτης και άλλων ισπανικών πόλεων αυτή τη στιγμή, γιατί απαντήσει υπάρχουν. Αυτή πιστεύω ότι είναι η σωστή κατεύθυνση και έτσι πρέπει να δουλέψουμε επικοδομητικά και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει δίκιο ο συνάδελφος Έρκας που μιλά για την ανάγκη επενδύσεων. και οι οργανώσεις εργοδοτών και οι οργανώσεις εργαζομένων και το κράτος θα πρέπει να συνεισφέρουν επενδύοντας στο μέλλον και στις θέσεις απασχόλησης για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και για την κατάρτιση και για την εκπαίδευση και για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Ένα σημαντικό θέμα και πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα αυτού του εγγράφου. Ε, χαίρομαι που αναφέρατε την ανάλυση του ΣΕΝΤΕΦΟΠ, γιατί είναι εξαιρετική η ανάλυση του ΣΕΝΤΕΦΟΠ που ανέφερε η συγκεκριτή του θέματος και υπάρχουν πολλές προτάσεις τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Είναι ένας φορέας που κάνει σημαντικό έργο και πρέπει και εμείς να χρησιμοποιούμε τα συμπεράσματά του. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μωράν και κυρία Λίν κατόπιν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Ρεγκίνα Μπάστος, για την εξαιρετική της δουλειά. Και την οποία μας παρουσίασε σήμερα. Όπως ακούστηκε, διορθώνει την οπτική γωνιά της Κομισιόν για να περάσουμε από τη flexicurity σε μια προβολή προς τη στρατηγική του 2020 η οποία ε, στρέφεται προς τις νέες δεξιότητες και τη νέα απασχόληση. Δεν Ρεγκίνα Μπάστος πολύ ε, σωστά υπογράμμισε τη μεγάλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, δηλαδή την μείωση της υφιστάμενης ανεργίας, κυρίως των νέων, αλλά και την ανανέωση των θέσεων εργασίας που ε, είναι, που συνδέονται σημαντικά με την ε, ηλικιακή ομάδα που ξεκίνησε με τα πολεμικά και που τώρα φτάνει στην ολοκλήρωση. Και βεβαίως έχουμε νέες ανάγκες των επιχειρήσεων και λόγω της παγκοσμιοποίησης. Μας προτείνε διάφορα πράγματα, στα οποία θα προσθέσω τρία που θεωρώ πολύ σημαντικά. Πρώτον, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ανεργίας και κυρίως της ανεργίας των νέων. Επ' αυτού μίλησε ε, ε, διαμακρόν και ο Αλεξάνδρος Σαρκάς. Σήμερα λέμε ότι οι χώρες που αντιστέκονται περισσότερο στην αύξηση ενεργείας των νέων είναι οι χώρες όπου το εκπαιδευτικό μοντέλο και κυρίως το η ακαδημαϊκή μόρφωση έρχεται σε επαφή με τις επιχειρήσεις για, ε, με τρόπους μαθητείας και θέλω να υπογραμμίσω ότι οι εναλλακτικές ε, παρακολουθήσεις και η μαθητεία δεν πρέπει να είναι μορφές ε, εκπαίδευσης που να απευθύνονται μόνο στους νέους που έχουν αποτύχει στο ακαδημαϊκό σύστημα. Είναι μορφές εκπαίδευσης εξαιρετικά αξιόλογες, εξίσου με, με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Ας πούμε, αναφέρομαι, ε, η εκπαίδευση των γιατρών και εδώ υπάρχουν γιατροί είναι τέτοια μορφής εκπαίδευση εναλλακτική ε, καθημαϊκή και άσκηση της, στην πράξη. Μάλλον, στην αρχική εκπαίδευση γίνεται ακαδημαϊκή, προσφέρεται ακαδημαϊκή μόρφωση και ε, μόρφωση στην επιχείρηση και όλες οι στατιστικές των 27 κρατών μελών δείχνουν ότι πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό το μοντέλο. Είναι και αυτό μια νέα αμφισβήτηση την οποία πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι εύκολο, είναι κάτι όμως που πρέπει να αντιμετωπίσουμε γιατί όπως συμβαίνει και στην Ισπανία, Αλεχάνδρο 44-45 για τους νέους 18-25 ετών που είναι ε, στην ανέργεια. Πρέπει να το μελετήσουμε αυτό το, αυτό το μοντέλο. Ένα δεύτερο σημείο επί του οποίου θέλω να παρέμβω είναι ότι δεν υπάρχει σε, σε καμία επιχείρηση μοντέλο κατάρτισης που να είναι αποτελεσματικό αν δεν υπάρχει ε, ε, επαγγελματική προσέγγιση από τον δάσκαλο, από τον εκπαιδευτή. Αν δηλαδή αυτός ε, ε, δεν γνωρίζει πώς να διδάξει, ε, Ε, ε, δεν θα είναι εξίσου αποτελεσματική αυτή η μέθοδος η οποία στηρίζεται στο να μάθει κάποιος με το να παρακολουθεί. Αλλά βεβαίως χρειάζεται και το διδακτικό στοιχείο. Και ε, τέλος, ποτέ δεν θα, δεν θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε εκπαιδευτές της επιχειρήσης και η κατάσταση στα 27 κράτη-μέλη μας επιβάλλει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα με επαγγελματικό τρόπο. Αυτή είναι η δεύτερη πρόταση που κάνω για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Και, ε, Ρεγκίνα, θέλω να κάνω και μια τρίτη πρόταση. New skills, new jobs λέμε, όλοι συμφωνούν. Όμως, αν θέλουμε να ανταποκριθούμε όπως προτείνεται και στην παράγραφο 9 να ανταποκριθούμε με τρόπο κατάλληλο που να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες που επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο οι πράσινες και περιβαλλοντικές θέσει εργασίες, είναι και αυτές, αλλά όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι θα πρέπει να κινητοποιηθούν, θα πρέπει να σκεφτούν τις νέες επαγγελματικές ανάγκες σε κάθε χώρο. Προτείνω λοιπόν η εργασία αυτή να γίνει με τρόπο σωστό και κατάλληλο ανά επαγγελματικό κλάδο ανά, αλλά και ανά επίπεδο προσόντων. Και, η Ευρώπη, προσόντων. και η Ευρώπη πρέπει να δείξει το δρόμο για αυτή τη νέα σύμβαση που πρέπει να συναυθεί ε, στους επαγγελματικούς κλάδους έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νέες αυτές ανάγκες. Αυτά είχα να πω ε, για να βοηθήσω να πετύχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Κυρία Λίν. Ευχαριστώ. Καταρχήν ζητώ συγγνώμη που δεν μπορούσε να παρευρεθεί, δεν να παρευρεθεί η κυρία Χάρκιν γιατί ε, ασθενή. Ε, για τη συγκεκριμένη έκθεση θέλω να πω ότι είναι καλή η έκθεση αυτή ε, για μια έκθεση της Επιτροπής την οποία θεωρώ επίσης καλή. Είναι σημαντικά τα θέματα της ε, μαθητείας ε, και είπατε κι εσείς, ε, η προηγούμενη ομιλήτρια, πόσο σημαντική είναι η μαθητεία. Αλλά δεν χρειάζεται μόνο μαθητεία και μετά να μην υπάρχει απολύτως τίποτα. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για κατάρτιση που θα οδηγήσει σε απασχόληση, όχι απλώς κατάρτιση που μετά δεν θα αποφέρει τίποτα στους καταρτιστέντες που θα παραμείνουν άνεργοι. Μετά όταν μιλάμε για τις δεξιότητες ε, θα πρέπει να ε, το επεκτείνουμε και σε κάποιες περιοχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει ίδια αναγνώριση προσόντων ε, και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άτομα που έρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο θέμα έχει σχέση με τη δουλειά του Τόμας Μαν για την ενεργό γύρανση και η Κίνγκα Γκόνς νομίζω ότι είχε κάνει μια τροπολογία ακριβώς ε, για την κατάρτιση ε, για άτομα που βρίσκονται στον τομέα της περίθαλψης. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και κάτι περισσότερο, πάντως σας ευχαριστώ που το έχετε ήδη συμπεριλάβει. Ο κύριος Σέρκα ανέφερε κάτι σε σχέση με την ευελιξία με ασφάλεια, flexicurity, και τα σημείωσα αυτά που είπε. Εσείς είπατε ότι δεν μπορεί η ευελιξία με ασφάλεια από μόνη τη να αποτελέσει ένα αντίδοτο στην κρίση. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να είναι το μοναδικό μέτρο. Πάντως χαίρομαι που αναφέρετε αυτό το σημείο σχετικά με την ευελιξία με ασφάλεια και μας ενδιαφέρουν όλοι οι πολίτες που ε, ε, είναι περισσότερο οριακοί όπως είναι οι ηλικιωμένοι, όπως είναι οι άνεργοι κλπ. Για την ε, ισότητα των φίλων χαίρομαι γιατί δεν ακολουθείτε την προσέγγιση που πολλές φορές ακολουθούμε στην Επιτροπή μας για τη συμφιλίωση ε, της οικογένειας και της επαγγελματικής ζωής, γιατί πολύ συχνά λέμε ότι αυτό θα ωφελήσει τις γυναίκες που θα τις φέρει στην αγορά εργασίας. Χαίρομαι γιατί λέτε ότι η συμφιλίωση εργασιακής και οικογενειακής ζωής θα φέρει περισσότερα άτομα και άνδρες και γυναίκες στην αγορά εργασίας. Τα θέματα της ε, φροντίδας των παιδιών μερικές φορές θα θεωρούμε θέματα που αφορούν τις γυναίκες, ενώ είναι θέματα που αφορούν τους γονείς και όχι μόνο τις γυναίκες και εσεί πολύ σωστά το έχετε θέσει, λέτε συμμετοχή, θα βελτιώσει τη συμμετοχή και των ανδρών και των γυναικών στην αγορά εργασία. Είναι πολύ καλή έκθεση και ξέρω ότι και η Μάριαν Χάρκιν θα έχει ως κοιόδηση συζητήτρια και εκείνη κάποια επιπλέον σχόλια από αυτή τη έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν, υπάρχει κάποιο άλλο που ζητάει το λόγο. Από ό,τι φαίνεται όχι. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Μήπως θα μπορούσε η Κομισιό να μας πει Πού βρισκόμαστε όσον αφορά την εφαρμογή αυτή τη πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή, στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ποιο σημείο βρίσκονται οι συζητήσει με τα κράτη-μέλη. Um, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε συντομία που βρισκόμαστε να αφορά την εφαρμογή. Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτή η πρωτοβουλία είναι ένα μέτρο το οποίο μας βοηθάει να πετύχουμε το στόχο του 77% και έχουμε τέσσερις προτεραιότητες, η λειτουργία της αγοράς εργασίας, δίνουμε μια, ένα νέο momentum στην Flexi Security, βελτιώνουμε τα προσόντα, την ποιότητα εργασίας και συνεισφέρουμε στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Υπάρχουν 31 δράσεις κλειδιά που συζητήθηκαν σε ένα κοινωνικό φόρουμ τριμερές το οποίο συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το FLEXSHIP σαν ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει να εντάξουμε στην προσπάθειά μας και τους κοινωνικούς εταίρους, κυρίως όσον αφορά τις πολιτικές του Flexi Security. Στις 10 με 11 Μαρτίου ε, συζητήθηκαν, έγινε αυτή η συνάντηση, μετά ε, τον ορισμό των τεσσάρων προτεραιοτήτων το συζητήσαμε περισσότερο την, το περιεχόμενο της μερισίας διάταξης. Ε, η συνάντηση αυτή θεωρήθηκε επιτυχής γιατί είχαμε ένα feedback και από τους κοινωνικούς εταίρους. Και αυτή η συνάντηση θα οργανώνεται σε αιτήσια βάση. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός που αφορά την Flex Security είναι μια διάσκεψη που θα μας επιτρέψει, μια σύνοδος τέλος πάντων που θα μας βοηθήσει ε, να συζητήσουμε το περιεχόμενο της ανακοίνωσης μια συνάντηση σύνοδος των stakeholders που θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο και ε, θα συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλοι οι stakeholders, τέλος πάντων, όλοι οι εμπλεκόμενοι. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή συγκυρία, θα είναι πολύ έγκυρη, η, η έκθεσή σας και θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική συνεισφορά στην όλη συζήτηση για την ε, περαιτέρω ανάπτυξη της έννοιας της ε, Flex Security η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού προετοιμάζει μία ανακοίνωση για την διαβίου εκπαίδευση που θα δημοσιευθεί σύντομα. Τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, δεν μπορώ να σας πω. Τέλος πάντων δεν μπορώ να σας πω ακριβή ημερομηνία, αλλά θα είναι σύντομα. Άλλες ε, είναι ε, ενεξελίξει για την επόμενη χρονιά. Υπάρχει το πανόραμα ευρωπαϊκών προσόντων, ευρωπαϊκό πανόραμα προσόντων. Όσον αφορά την ε, ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ε, προτείνουμε μία σειρά αρχών, κατευθυντηρίων αρχών, που θα διέπουν την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, κάτι που είχαμε προβλέψει εδώ και καιρό αλλά θα το δημοσιευτεί του χρόνου κάποια στιγμή. Αυτά με λίγα λόγια που βρισκόμασταν και περιμένουμε με ανυπομονησία τη συνεισφορά σα δηλαδή την έκθεσή σας. Ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις σας και θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, κυρία Μπάστος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Οφείλω να ομολογήσω ότι ε, εκτίμησα ιδιαίτερα τη συνεισφορά όλων των συναδέλφων που συμμετείχαν σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα, είναι συμβολικό θα έλεγα σε αυτή την περίοδο που διανύουμε τώρα που πρέπει η Ευρώπη να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες προκλήσεις που ε, δημιούργησε η κρίση. Ε, οι συνεισφορές ήταν πάρα πολύ σημαντικές πιστεύω και συγκεκριμένες. Δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια κάποια ε, δυναμική ανάπτυξη ε, που θα οδηγήσει στην αύξηση της απασχόλησης ε, με την βοήθεια των επιχειρήσεων που θα δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και θα δίνουμε και την δυνατότητα στους πολίτες, θα δίνουμε μεγαλύτερες δυνατότητες αν θέλετε στους πολίτες, εκπαιδεύοντας τους να αποκτήσουν μια αξιοπρεπή δουλειά και ε, σε, προχωρημένο, σε μια προχωρημένη ηλικία. Όλα αυτά πιστεύω ότι εντάσσονται και με την κουλτούρα μας και με το κοινωνικό μας μοντέλο, αλλά και ε, τονίζουν την θέλησή μας να είμαστε στο προσκήνιο και να καινοτομούμε στον, ε, στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομίας. θα πρέπει να δημιουργηθούν βέβαια και οι απαραίτητες συνθήκες που θα εξασφαλίσουν και την ευημερία των πολιτών μας. Υπάρχει βέβαια και αυτό το, ε, το κουδούνι, τον κουδούνι κινδύνου που θα πρέπει να κρούσουμε για την flex security. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τομέα αυτό θέλουμε να ακολουθήσουμε τον δυναμισμό και της αγοράς εργασίας που δεν μπορεί να μείνει στάσιμη και ε, εξελίσσεται συνέχεια και εμείς θα πρέπει όντως να δώσουμε ε, μία απάντηση σε αυτή την ε, πραγματικότητα η οποία αλλάζει καθημερινά. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι ιδιαιτερότητες ε, κάθε περιοχής, ε, κάθε χώρας, άρα δεν μπορεί να έχουμε μια ενιαία απάντηση. Επίσης ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το θέμα των εκπαιδευτών αν θέλετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε την ζήτηση και την προσφορά θέσεων απασχόλησης. Όλοι, όλοι οι συνάδελφοι είπαν ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει με τις ε, τροπολογίες της να μας προετοιμάσει για το επόμενο στάδιο που αποτελεί και κίνητρο αλλά και πρόκληση για να λύσουμε ε, θέματα πάρα πολύ δύσκολα όπως προς χάρη η νεανική ανεργία, η ανεργία των νέων. Ε, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής αναφέρθηκε στο, στη συνάντηση αυτή που θα ασχοληθεί με τα θέματα της Flexus Security. Περιμένω με ανυπομονησία το, το γεγονός αυτό, την εκδήλωση αυτή. Λοιπόν, στην ακρόαση της 15ης Ιουνίου σας περιμένω. Ελπίζω να είστε πολλοί και να κάνετε επικοδομητικά σχόλια, σαν και αυτά που κάνετε και εδώ. Merci. Ευχαριστώ την αγαπητή εισηγήτρια. Πράγματι θα οργανώσουμε την ακρόαση στις 15 Ιουνίου με τους ε, κοινωνικούς εταίρους. Συνειδητοποιώ όμως ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών που ορίσαμε είναι με προηγουμένη, ε, είναι πιο κοντά μας, 6, 7 Ιουνίου θα μελετήσουμε στις 12 και 13 Ιουνίου. Και βεβαίως η αυτά που θα ακούσουμε από τις 15 Ιουνίου θα πρέπει να ενσωματωθούν μέσω προφορικών τροπολογιών κτλ. κτλ. Θα τελειώσουμε τώρα με αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης και προχωράμε στο σημείο 14, οπότε θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο Τράιεν Ουγγουρεανού, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την έκθεσή του για της οποίας είμαστε ε, υπεύθυνοι ε, στην ουσία προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε τις συμβιβαστικές τροπολογίες που συντάξατε επί τη βάση των 157 τροπολογιών που δεχτήκατε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σωστά τα λέτε. Αυτή η έκθεση αφορά την ενθάρρυνση της κινητικότητας των εργαζομένων, όπως είπατε. Αυτή είναι η ουσία της έκθεσης. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και οι συνάδελφοι με τις επικοδομητικές παρατηρήσεις και τροπολογίες τους και τους είμαι ευγνώμων για την επικοδομητική του στάση. Θα προσπαθήσω να σκιαγραφίσω τις συμβαστικές λύσεις τις οποίες έχουμε καταλήξει. Ξεκινάω με τις πρώτες συμβαστικές λύσεις που έχουν ως στόχο να ασχοληθούμε με τα θέματα που μέχρι τώρα δεν μας έχουν απασχολήσει επαρκώς όσον αφορά την κινητικότητα θέλω να αναφέρω την έλλειψη συγκεκριμένων μέτρων για την υποστήριξη της κινητικότητας. Αυτό είναι μια διατύπωση που έχουμε πάρει από την κοινοποίηση της Επιτροπής. Είναι σωστή αυτή η θέση του Κοινοβουλίου και δίνουμε το μήνυμα ότι πρέπει να λάβουμε δράση και συγκεκριμένα μέτρα για τις δύο πρώτες συμβιβαστικέ λύσεις, την Α και Β, θέλω ακόμη να πω ότι υπάρχει ανάγκη να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα των ατόμων που αναζητούν νέες αγορές εργασίας και που επομένως μετακινούνται. Εδώ θα ήθελα να τονίσω και το δικαίωμα ψήφου γιατί το δικαίωμα του εκλέγην είναι ένα σημαντικό δικαίωμα. Οι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορούν να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μία ένωση και να μην εμποδίζεται κάποιο πολιτικό τους δικαίωμα λόγω της μετακίνησής τους. Ακόμη και αν πρόκειται για ένα δικαίωμα το οποίο αφορά τη χώρα προέλευσής τους ενώ βρίσκονται σε άλλη χώρα. Περνάω στην τρίτη συμβιβαστική λύση, συμβιβαστική τροπολογία C, που είναι αυτή που συζητήσαμε περισσότερο νομίζω. Τη συζήτησα με τους συναδέλφους και εδώ υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να αναφέρουμε ιδιαίτερα. Σε αυτή την τρίτη συμβιβαστική τροπολογία λοιπόν, καταρχήν πρόκειται για την ισορροπία μεταξύ των εθνικών νομικών πλαισίων για την απασχόληση. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθετικών πλαισίων. Η αρχή της συλλογικής σύμβασης εργασίας θα πρέπει να επικρατήσει και θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση για δίκαιους κανόνες ανταγωνισμού. Κατάργηση των φραγμών που θα μπορούσαν να εμποδίζουν την πρόσβαση στην απασχόληση για τους μετακινούμενους εργαζομένους είναι κάτι το οποίο είναι εγγυημένο όταν έχουμε θεσπίσει ότι μια δουλειά χρειάζεται ένα συγκεκριμένο επίπεδο δεξιοτήτων ή γνώσεων. Και αυτό το επίπεδο θα πρέπει να είναι δίκαιο προς όλους, δηλαδή ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης του εργαζομένου, θα πρέπει να δίνουμε σημασία στο επίπεδο των προσόντων. Και όσον αφορά την ίδια τροπολογία, την τρίτη συμβιβαστική τροπολογία, έχουμε προσθέσει ε, όχι μόνο το κοινωνικό ντάμπινγκ αλλά και το μισθολογικό ντάμπινγκ. Στην επόμενη τέταρτη συμβαστική τροπολογία, Μιλάμε για τα δικαιώματα των μετακινούμενων εργαζομένων ε, για την, στην υγειονομική περίθαλψη. Για να διευκολύνει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η χώρα υποδοχής θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα αρχεία των εργαζομένων και δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται η πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία. Λάβαμε υπόψη μας ότι τα συστήματα υγείας των διαφόρων χωρών διαφέρουν και δεν είναι ρόλο της παρούσας έκθεσης να ζητήσει την εναρμόνιση των συστημάτων υγείας. Ούτε ζητάμε να είναι ομοιόμορφα τα συστήματα υγείας στο μέλλον, αλλά θέλουμε να υπάρχει πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους. Περνάω στην πέμπτη συμβιβαστική τροπολογία. Αυτή η σεβαστική τροπολογία προσπαθεί ε, να δείξει ότι θέλουμε ένα θετικό αντίκτυπο για την αγορά εργασίας. Δηλαδή, να σας πω ποιο είναι το σκεπτικό, ότι η μετανάστευση είναι κάτι το καλό, είναι κάτι το ευεργετικό για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες που τονίζουν και τα θετικά στοιχεία και τα μειονεκτήματα της μετανάστευσης. για την οικονομία δηλαδή των κρατών μελών. Και πιστεύω ότι πρέπει να τονίσουμε τα πλεονεκτήματα, αλλά να δώσουμε και σημασία και στα μειονεκτήματα τα οποία μερικές φορές δεν λαμβάνονται υπόψη. Αν εξισορροπήσουμε λοιπόν τα θετικά με τα αρνητικά σημεία, θα μπορέσει να προκύψει μια πιο ακριβής εικόνα, ούτω ώστε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι είναι μεγαλύτερα τα πλεονεκτήματα από τα μειονεκτήματα. Οι επόμενες δύο συμβιβαστικές τροπολογίες, η F και η G, εξετάζουν τη σημασία της πρόσβασης στην πληροφόρηση μέσω του δικτύου EURES και εδώ το θέμα είναι η ποιότητα των δεδομένων που προσφέρονται στους μετακινούμενους εργαζομένους. Η συνδεστική τροπολογία H, ήτα, δεν είναι καθόλου προβληματική. Απλώς εδώ δηλώνουμε ότι η κινητικότητα δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι είναι μονοπόλιο των νέων. Η αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται και την πρακτική εμπειρία την οποία συσσωρεύει κανείς μέσω των πολλών ετών υπηρεσίας και η κινητικότητα της εργασίας θα πρέπει να αφορά όλους, όλες τις ε, ηλικιακές ομάδες και όλες τις κατηγορίες. Η επόμενη συμβαστική τροπολογία, η I, Ι, εξετάζει τα εκπαιδευτικά συστήματα και εδώ ε, λέμε ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ακόμη τονίζεται ότι έχει σημασία η αναγνώριση των διπλωμάτων και η αναγνώριση των προσόντων για τα κλειστά επαγγέλματα. Γιατί αν θέλουμε να επιτύχουμε πραγματική οικονομική σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητο αυτά τα σημεία. Στην επόμενη συμβαστική τροπολογία, την J, ασχολούμαστε με ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα, το θέμα της χρήσης ξένων γλωσσών. που και στο παρελθόν αλλά και ακόμη έχει τύχει να οδηγεί σε καταχρηστικές πρακτικές έναντι των μετακινουμένων εργαζομένων, κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Η συμβαστική τροπολογία λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται την ε, μετανάστευση. Επομένως αποτελεί ένα σημείο αφετηρίας αυτή η συμβαστική τροπολογία για την ε, όλη γνωμοδότηση. Και εδώ διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό των μεταναστών είναι ακόμη χαμηλό σαν μέσο όρο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, η συνδεσική τροπολογία L ασχολείται με την αναγνώριση των διπλωμάτων των επαγγελματικών προσόντων ούτως ώστε να ανταποκρινόμαστε σωστά στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Προσπάθησα να συνοψίσω τις συμβαστικές τροπολογίες και δεν έχω άλλα σχόλια προς το παρόν. Ευχαριστώ. Euh, Ωραία. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση hm? και θα δώσω το λόγο στις συναδέλφους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανα και για την ε, έκθεση αλλά και για τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα ε, ικανοποιεί όλες τις πολιτικές ομάδες. Χαίρομαι που καταλήξαμε σε συμφωνία ε, για τις συμβαστικές τροπολογίες τροπολογίες που αφορούσαν και τις συνθήκες εργασίας για την πρόληψη του κοινωνικού ντάμπινγκ και καταφέραμε να συμφωνήσουμε ακόμα και για την ανάγκη αναγνώρισης των, ε, της αμοιβαίας των, κοινωνικών προσω... των επαγγελματικών προσόντων και των διπλωμάτων. Ε, βέβαια, είναι κρίμα γιατί δεν ε, καταλήξαμε σε συμφωνία για όλα τα θέματα παραδείγματος χάρη ε, για τους μισθούς παραδείγματος χάρη ή για την συμμετοχή σε συνδικάτα. Αυτά είναι πάρα πολύ βασικά θέματα πιστεύω για να μπορούμε να προωθήσουμε την ε, μετακίνηση των εργαζομένων και για να μπορούν οι εργαζόμενοι να ε, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ψηφίσουμε και, και σε άλλες επιτροπές για το κείμενο αυτό και ελπίζω ότι αυτή το αποτέλεσμα της εργασίας των άλλων ε, επιτροπών θα βοηθήσει και θα συνεισφέρει ε, στις εργασίες μας. Ε, κυρία Λίνα. Ευχαριστώ. Η Μάριν Χάρκιν δεν μπορεί ε, να παρευρεθεί γιατί ασθενεί. Ενώ είναι βέβαια η σκιώδης εισηγήτρια και μου ζήτησε να διαβάσω μια σύντο, ένα σύντομο κείμενο. Είπε ότι θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά που έκανε και τη σύνταξη των συμβασικών τροπολογιών. Με τα χαρά διαπίστωσε ότι πολλέ από τι διαπραγμα... από λήφθηκαν υπόψη, της, ε, υπόψη κατά τη διάρκεια τη προετοιμασία και ε, μέχρι τώρα είναι πολύ απολύτω ικανοποιημένη. Όμως προσβλέπει τη συνεργασία με τον εισηγητή στην επόμενη, στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων. Άρα, προφανώς υπάρχουν ένα-δυο σημεία που θα θέλει να διαπραγματευτεί όταν επιστρέψει από όταν, και όταν έχει γίνει κάποια καλά δηλαδή. Ευχαριστώ κύριος Κρίστενσεν. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή ο οποίος κατάφερε να πετύχει μια σωστή ισορροπία. Έτσι ε, παραμένουν κάποια δικαιώματα στις συλλογικές συμβάσεις ή ε, στην νομοθεσία της χώρας προέλευσης. Ζήτησα το λόγο διότι ε, θέλω να σχολιάσω τον ε, συμβιβασμό B και τον συμβιβασμό F με επί τη βάση συγκεκριμένων παραδειγμάτων από τη Δανία. Διαπιστώσαμε ότι οι εργαζόμενοι, οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα που θα τους επιτρέψουν να έχουν πρόσβαση σε νοσηλεία και βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση ανθρώπου που ε, η δαπάνη έφτανε τα 2 εκατομμύρια κορώνες και δεν ξέρανε ποιος να τις καταβάλει, ποιος να τις πληρώσει. Υπάρχει ε, ένα έγγραφο, το ε, έγγραφο ένα που προβλέπει ότι ε, ο εργοδότης αναλαμβάνει την ευθύνη. Άρα πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Αυτός ο οποίος μετακινείται οπουδήποτε στην Ευρώπη θα έχει μία εγγύηση ότι μπορεί να νοσηλευθεί σε ένα νοσοκομείο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σας ευχαριστώ πολύ. Έλειψα για λίγο γιατί ήμουν στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και έπρεπε να είμαι εκεί σε κάποια ψηφοφορία. Ε, είχα μια ερώτηση για την τροπολογία 104. Γιατί ήδη πέρυσι όταν έγιναν οι διαπραγματεύσεις για το τι γίνεται με την ελεύθερη διακίνηση από 1η Μαΐου είχα κάνει μια ερώτηση τότε προς την Επιτροπή και τους είχα ζητήσει να κάνει μια μελέτη. Ποια είναι η θέση του εισηγητού για την τροπολογία 104. Ε, τι θα πρέπει να αναμένουμε για την εξέλιξη των αγορών εργασίας, ε, τι γίνεται με τις μεταβατικές ρυθμίσεις. Δεν έχουμε πια δυνατότητα στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, να παρατείνουμε τη μεταβατική περίοδο και σωστά δεν έχουμε πλέον, αλλά ε, ποιες είναι οι επιπτώσεις της ελεύθερης διακίνησης. Ε, στη Γερμανία σίγουρα χρειαζόμαστε ε, εργαζόμενους ε, και χρειαζόμαστε και νέους οι οποίοι χρειάζονται κατάρτιση. Είναι πολλά λοιπόν τα σημεία τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, και γι' αυτό χρειάζεται μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επιπτώσεις και θα έπρεπε μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 να την έχουμε αυτή τη μελέτη. Εγώ τουλάχιστον αυτό ζητάω. Εκτό αν ο εισηγητή πιστεύει ότι δεν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να ακούσω την ε, γνώμη σα επ' αυτού. Δεν λέω να κάνουμε μια μελέτη ε, ε, απλώς και μόνο για να έχουμε μια μελέτη, αλλά γιατί θέλουμε να υπάρχει μια πρόγνωση, να ξέρουμε τι να περιμένουμε και να ξέρουμε ότι είναι θετικό το να έχουμε ε, ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και να μην κλείνουμε τα σύνορά μας ε, στους μετακινούμενους εργαζόμενους. Αυτή η μελέτη εγώ θεωρώ ότι είναι χρήσιμη. Εσείς τι γνώμη έχετε. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Άλλες ερωτήσεις. Πριν δώσω και πάλι το λόγο στον εισηγητή, δεν συμμετέσχω στην ε, κατάτηση των τροπολογιών αλλά λαμβάνοντα υπόψη τα όσα συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τομείς και λαμβάνοντα υπόψη και τις απειλές προς τον μηχανισμό Schengen, το θέμα της κινητικότητας των εργαζομένων χωρίς να αναφέρεται καθόλου αυτή η διάσταση που σαφώς έχει καθοριστική επίπτωση στην κινητικότητα των εργαζομένων θα ήταν τουλάχιστον περίεργο το να μην το αναφέρουμε καθόλου. Ε, κάνω αυτή την παρατήρηση και την αφήνω στη σοφία του εισηγητού, ε, έστω και μέσω μιας προφορικής τροπολογίας, να κάνει μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Μιλάμε για τα δικαιώματα ψήφου των ε, εργαζομένων κλπ. Ε, ε, αλλά δεν μπορούμε να γνωρούμε ότι παράλληλα κάποια κράτη-μέλη κλείνουν τα σύνορά τους ε, δεν προτείνω να κάνουμε μια έκθεση που δεν θα είναι προσαρμοσμένη στην παρούσα κατάσταση στην Ευρώπη, ξέρω ότι πρέπει να ε, ε, απαντήσουμε σε μια ανακοίνωση της Επιτροπής που έχει συγκεκριμένο αντικείμενο και ε, είναι μια ανακοίνωση από πέρυσι τον Ιούλιο. Αλλά δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μας το πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνουν όλα αυτά. Υπάρχουν λοιπόν κάποιε παρατηρήσει που νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ που θέτετε τέτοια θέματα, που είναι θέματα αρχής. Θα προσπαθήσω ένα-ένα να τα πιάσω τα διάφορα θέματα. Η κυρία Βλίνκεβιτσούτε ανέφερε το πρόβλημα του δικαιώματος ένταξης σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και το δικαίωμα απεργίας. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να επισημάνουμε το α ή το β δικαίωμα ε, ή κάποια κατηγορία δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να μιλάμε γενικά για θεμελιώδη δικαιώματα. Να μην αναφέρουμε συγκεκριμένα δικαιώματα όπως το δικαίωμα ε, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή το δικαίωμα απεργίας. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις εκ μέρους της κυρίας Χάρκιν. Να έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα και συμφωνώ και για τα θέματα για τα προβλήματα ε, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Κρίστανσεν, ότι πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Ε, για την παρατήρηση του συναδέλφου κυρίου Τόμας Μαν σχετικά με την κατάρτιση μιας μελέτης. Εγώ θα έλεγα ενδεχομένως μια νέα μελέτη για τις επιπτώσεις της μετακίνησης των εργαζομένων στην ε, αγορά εργασίας. Διότι ήδη έχουμε μελέτες και ήδη υπάρχουν και προηγούμενα και θα έλεγα μάλιστα ότι ήδη γνωρίζουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν συμβεί και συνεχίζουν να συμβαίνουν όταν μπαίνουν ε, εργαζόμενοι στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας φέρω το παράδειγμα του τι συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο. όπου υπήρχε μεγάλος φόβος ότι πρόκειται να ε, έρθουν κύματα Πολωνών εργαζομένων που θα κατέκλυζαν τα Βρετανικά νησιά περίμεναν 300.000 εργαζομένους στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα. Και τελικά τι συνέβη. 30.000 ήρθαν και όχι 300.000 εργαζόμενοι. Δεν δημιουργήθηκε λοιπόν κοινωνικό πρόβλημα. Δημιουργήθηκαν πολλά ζητήματα στον τύπο, αλλά κοινωνικό πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε. Ως Γενική Αρχή λοιπόν γνωρίζουμε ότι η μετανάστευση είναι κάτι το θετικό. Χωρίς βέβαια να ισχυριζόμαστε ότι δεν είναι προβληματικό. Προβλήματα υπάρχουν. Και εδώ συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα μειονεκτήματα τις αρνητικέ επιπτώσεις είπατε. Θα έλεγα τα μειονεκτήματα για να μην πούμε αρνητικέ επιπτώσεις. Εάν υπάρχουν προβλήματα από την μετανάστευση εργαζομένων, ιδίως όταν μιλάμε για εργαζομένους από την Βουλγαρία και τη Ρουμανία που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα μετακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως είναι περισσότερο πρόβλημα ε, του πώς ε, το εκλαμβάνουμε, γιατί είναι θέματα τα οποία εκμεταλλεύεται πολιτικά η ακροδεξιά. Και η ουσία της έκθεσης αυτής είναι να ενθαρρύνουμε την νόμιμη μετανάστευση και όχι να περιορίσουμε τη μετανάστευση. Δεν αμφισβητούμε τα θετικά σημεία της μετανάστευσης, θέλουμε να τη διευκολύνουμε. Και η Πρόεδρος ε, έθεσε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Να το πω με άλλα λόγια. Είπατε πώς μπορούμε να μιλάμε για τη μετανάστευση στην Ευρώπη όταν λίγο πολύ δεν υπάρχει το Σέγγεν πλέον. ευτυχώς ισχύει ακόμη η Συμφωνία Σέγγεν. Ναι, συμφωνούμε από αυτού. Ευτυχώς ισχύει ακόμη. Και τα θέματα που αφορούν τη μετανάστευση δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με πολιτικές βλέψεις. Κάποιες χώρες στην Ευρώπη είτε λαμβάνουν είτε απειλούν ότι θα λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της μετακίνησης εργαζομένων. Και το θέμα αυτό το συζήτησα ήδη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που κάναμε. Και εδώ συμφωνούμε απολύτως ότι τέτοια μέτρα θα ήταν αντίθετα προς την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θα πρέπει ε, να υπάρξει αντίσταση σε τέτοια μέτρα ή να ανακληθούν αν υπάρξουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την τόσο λεπτομερή απάντηση. Ε, θα ψηφίσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες στην επόμενη συνάντησή μας, δηλαδή κάποια στιγμή 15-16 Ιουνίου, μάλλον στις 16, 16 Ιουνίου, σύμφωνα με την πρακτική μας και Μέχρι τότε νομίζω ότι θα έχουμε πάρει... Υπάρχει γνωμοδότηση επιτροπής. Λοιπόν, μέχρι τότε θα έχουμε εξετάσει και τις ε, γνωμοδοτήσεις ε, των ε, Επιτροπών Γυναικών και Ελευθεριών. Λοιπόν, τελειώσαμε με την σημερινή μας εργασία. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 9. Ευχαριστώ.